Okay. Well, good afternoon, everybody. Um, I'm sorry about the absence Είχαμε μία σειρά συναντήσεων. Γι' αυτό θα ήθελα όλοι να προσθέσουν εδώ το σύντομότερο. Ξέρω ότι ο Υπουργός πρέπει να φύγει σε μία ώρα περίπου και έχει πολλά και σημαντικά να μας πει. Θα θέλαμε να του υποβάλουμε και ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την φιλοξενία σας και γιατί οργανώσατε μία σειρά συναντήσεων όταν σας συναντήσαμε τον Απρίλιο. Εν ώψη της Προεδρίας γνωρίσαμε συναδέλφους σας που ασχολούνται με πολιτικά θέματα. Θέλουμε να οικοδομήσουμε σχέσεις με τις ε, προεδρίες, με τις επερχόμενες και τις προηγούμενες μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών μας ενδιαφέρει να έχουμε καλές και ποιοτικέ σχέσεις πριν από την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν για πρώτη φορά με μεγάλη χαρά ο ρόλος σας είναι ζωτικής σημασίας. Γνωρίζουμε ότι τον αναλαμβάνετε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ασχολείστε με θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και τουρισμού. Πολύ πτυχό το έργο σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε και στη συνέχεια θα σας υποβάλουμε ερωτήσεις σε σχέση με το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, και για τα καλά σας λόγια. Ε, κυρία Αντιπρόεδρος, ε, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, η σημερινή παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα ενώπιον της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ αποτελεί η συνέχεια μια καθιερωμένη πρακτική να ενημερώνεστε από την Προεδρία του Συμβουλίου για τις προτεραιότητε και δράσει που αναλαμβάνει να προωθήσει κατά τη διάρκεια τη εξάμεινη ιδία τη στα θέματα της εσωτερικής αγοράς, των καταναλωτών και τη τεχνική εναρμόνισης. Όμως, πολύ πέραν τη ανταπόκριση μου σε καθιερωμένε πρακτικέ, η εδώ παρουσία μου είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού μου απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατικότερη, να πλησιάσει περισσότερο και να αφουγκράζεται καλύτερα τους πολίτες της. Άλλωστε, κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι για μια καλύτερη Ευρώπη, πρώτα και κύρια για τους πολίτες της. Από την έναξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουν διευρυθεί οι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω συνομοθέτη με το Συμβούλιο. εκπροσωπώντα εδώ, εδώ την Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνουμε την ετοιμότητά μα να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε με επιτυχία του φακέλου που θα διαχειριστούμε το δεύτερο εξάμεινο του 2012 στου τομεί τη αρμοδιότητά μα. Στην αρχική μου αυτή παρέμβαση συνοπτικά θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας πολιτικές και τα επιμέρους θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξι μήνες όπως συμφωνήθηκα στο πλαίσιο του τρίου της Προεδρίας. Με αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Πολωνική όσο και τη Δανική Προεδρία για τη συνεργασία που αναπτύξαμε όλη αυτή την περίοδο αλλά και να τους συγχαρώ για την επιτυχή διαχείριση σημαντικών φαγγέλων που ανέλαβα. Έργο βέβαια που έχει παραχθεί με τη σημαντική συμβολή και συνεργασία τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών, αλλά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, μέλη τη Επιτροπή, σα χαίρω για αυτό σα το έργο. Κυρίε και κύριοι, οι στόχοι τη Κυπριακή Προεδρία για την Εσωτερική Αγωνά κινούνται σε δύο κύριου άξονε. Πρώτον, την πρόθεση και όπου είναι δυνατό ολοκλήρωση τη διαδικασία υιοθέτηση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσει τη υφιστάμενης πράξη για την ενιαία αγορά 1. Οι προτάσεις βέβαια για τις οποίες εκκρεμεί ακόμα η έγκριση είναι πολλέ, παρά τις ουσιαστικέ προσπάθειες που κατάβαλα οι δύο προηγούμενε Προεδρίες τη Πολωνία και της Δανία. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι με τη στενή συνεργασία τόσο με τους εταίρους μας στο Συμβούλιο, όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής πρόοδου. Άλλωστε, ο στόχος είναι κοινό και δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην ανάπτυξη, η τόνωση της απασχόλησης και η δημιουργία συνθηκών διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Δεύτερο, τη δρομολόγηση νέων δράσεων της πράξης για την ενιαία αγορά 2. Αναμένουμε την έγκαιρη έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένω ότι αυτό θα γίνει ε, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο προκειμένου να καταστεί δυνατή η ετοιμασία συμπερασμάτων από την Κυπριακή Προεδρία τα οποία θα τεθούν για έγκριση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου. Παράλληλα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, η Κυπριακή Προεδρία θα διοργανώσει στις 20 Οκτωβρίου ειδικό συνέδριο στη Λευκοσία με πρώτη στο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο για τα επιτεύγματα αλλά και τις δυσκολίες και τις προκλήσεις για το μέλλον. Όσον αφορά στις επιμέρους προτεραιότητες μας που εντάσσονται στην πράξη ενιαίας αγοράς επιτρέψτε μου να επεκταθεί λίγο στο θέμα των δημόσιων συμβάσεων. Κύριος στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η θεσμοθέτηση ενός απλοποιημένου, ευέλικτου και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα μειώνει το διοικητικό άχθος, θα παρέχει νομική βεβαιότητα και θα υποστηρίζει αφενός την εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, αηφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως εξάλλου είναι και η στρατηγική Ευρώπη 2020, και αφετέρου την πλέον αποδοτική χρήση των δημοσίων πόρων. Η εισαγωγή του μοντέλου εργασίας που εισήγαγε η Ιδανική Προεδρία, την προσέγγιση δηλαδή κατά σύμπλεγμα διατάξεων, cluster approach, ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό. Υιοθετούμε την πρακτική αυτή και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση το ίδιο μοντέλο. Πρόθεσή μας ως Κυπριακή Προεδρία είναι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια συνεργαζόμενη με την Επιτροπή σας όπως και με τα υπόλοιπα αρμόδια όργανα της Ένωσης προς επίδευξη τελικής συμφωνίας για δύο προτάσεις οδηγιών, την κλασική και της κοινή ωφελία μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, η επιδίωξή μα είναι οι κανόνες που θα υιοθετηθούν να διασφαλίζουν Πρώτον, την απλοποίηση και την αύξηση της ευελιξίας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με την προσέγγιση εργαλειοθήκης, των εξυγχρονισμών των διατάξεων και την προώθηση των ηλεκτρονικών συμβάσεων. Δεύτερον, τη στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων και την ανταπόκρισή τους στις νέες προκλήσεις με την επίτευξη της βέλτιστη προσλαμβανόμενης σχέσης ποιότητας τιμής την εισαγωγή του κόστου διαρκείας ζωής, την επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις του κοινωνικού, εργατικού και περιβαλλοντικού δικαίου και την πρόθεση της καινοτομίας. Τρίτον, την καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά με την απλοποίηση των υποχρεώσεων εγγραφής τεκμηρίωσης, την αποδοχή προσωπικών δηλώσεων ως προκαταρκτικά μέσα απόδειξης και τον περιορισμό των απαιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής. Τέταρτον, τις ορθές διαδικασίες με την αντιμετώπιση των επισφαλών επιχειρηματικών πρακτικών όπω η σύγκρουση συμφερόντων, η ευνοκρατία και η διαφθορά. Πέπτον, την καλύτερη διακυβέρνηση με τη διοικητική συνεργασία, τη δημιουργία και εκμετάλλευση κέντρων γνώσεων και την αποτελεσματική εποπτεία από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά στην πρόταση οδηγία για τι συμβάσει παραχώρηση, θεωρούμε ότι μια απλοποιημένη μορφή οδηγία με περιορισμένου κανόνε που θα διασφαλίζουν τι αρχέ της διαφάνεια, τη ίση μεταχείρισης και τη μη διάκρισης θα συμβάλλει στην κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαψη και τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή. Θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την επίτευξη συμφωνία. Εξίσου σημαντικό θέμα είναι και αυτό των επαγγελματικών προσόντων. Ο εξυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι υψή τη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη πράξη τη γενναία αγορά καθώ και για την Κυπριακή Προεδρία. Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να διευκολυνθεί η εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να καλύπτονται τυχόν ελλείψεις θέσεων εργασίας με τα συνεπακόλουθα ωφέλη για την αγορά εργασίας, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενδυνάμωση τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η απλοποίηση των κανόνων για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον καταστεί επίγουσα ανάγκη όπω και ενδυνάμωση τη συνεργασία και αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προωθήσει την πρόταση στον πλαίσιο των εργασιών τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει επαφέ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιδευθούν οι απαραίτητε συγκλήσει και στα δύο σώματα. Η πρόταση για την αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο η Κυπριακή Προεδρία ευελπιστεί ότι οι τριλόγοι που θα αρχίσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στεφθούν με επιτυχία και η ολοκλήρωση τη διαδικασία, η υιοθέτηση τη πρόταση θα καταστεί δυνατή πριν το τέλο του χρόνου. Όσον αφορά τα θέματα των καταναλωτών, η Κυπριακή Προεδρία θα αναλάβει θέματα που εμπίπτουν στι 12 δράσει για την πράξη για την ενιαία αγορά και που αποτελούν προτεραιότητα για όλους μας. Είναι πιστεύω αναγκαίο να θέσουμε τον πολίτη στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς με απότερο σκοπό να απολαμβάνουν οι πολίτες όλα τα ωφέλη της. Οι καταναλωτές διεκδικώντας ποικιλία, ποιότητα και αξιοπιστία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όπως και της Ένωσης εν γέννη. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι όπως οι πολίτες να είναι καλά προστατευμένοι με πιστή εφαρμογή δικαιωμάτων για τα οποία είναι καλά ενημερωμένοι. Όπως μας είναι άλλωστε γνωστό, οι καταναλωτικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 56% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επομένω προφανές ότι ένα περιβάλλον στο οποίο οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και έχουν εύκολη πρόσβαση στην έννομη προστασία είναι απολύτως απαραίτητο. Σε αυτό το πλαίσιο θα εργαστούμε για την ολοκλήρωση της πρότασης οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, την ATR, και της πρότασης κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, OTR. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον κύριο Χάκου, τον πρόεδρο της Επιτροπής και όλη την Επιτροπή για την άμεση ανταπόκριση ε, να συζητήσουν και να ψηφίσουν ε, τις συζητήσεις ε, που αφορούν την οδηγία και τον κανονισμό που μας δίνει τη δυνατότητα στο επόμενο χρονικό διάστημα να εργαστούμε συλλογικά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έγκριση και την ψήφιση της οδηγίας και του κανονισμού πριν από το τέλος του 2012. Στο κεφάλαιο αυτό και πέρα από την πράξη για την ενιαία αγορά, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει και θα στοχεύσει να ολοκληρώσει την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα καταναλωτών 2014-2020. ύψιστη προτεραιότητα για την Προεδρία μας αποτελεί επίσης η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προϊόντων. Ω εκ τούτου θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για εξέβραση συμβαστική συμφωνία όσον αφορά τη δέσμη των εννιά νομοθετικών προτάσεων που ευθυγραμμίζουν την υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Η Κυπριακή Προεδρία έχει ως στόχο να συμπληρώσει την εξέταση του φακέλου στην ομάδα εργασία και αφού συνεργαστεί επικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτύχει την υιοθέτηση του πακέτου σε πρώτη ανάγνωση οι προσπάθειες παροχής βελτιωμένων νομοθεσιών που ενισχύουν την ασφάλεια και ταυτόχρονα προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα ενισχυθούν μέσα από την επιδίωξή μας για ολοκλήρωση του φακέλου που αφορά την οδηγία για τα σκάφη αναψυχής. Η υιοθέτηση αυτή τη οδηγία θα εξασφαλίσει ισότιμου όρου κανονιστικών ρυθμίσεων με του κύριου εμπορικού εταίρου, καθώ και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σκαφών αναψυχής. Παρότι οι εργασίες για το συγκεκριμένο φάκελο βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, έχουμε τις καλύτερες ενδείξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν τα περιθώρια για επίδεξη συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχο της Κυπριακής Προεδρίας είναι να συνδράμει επικοδομητικά στην εξέλιξη του φακέλου. Όσον αφορά τους δύο κανονισμούς σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα Φαίνεται ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά στην εξέβρεση μιας συμβαστική λύση. Η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να συνδράμει επικοδομητικά για να επιτύχει την ολοκλήρωση των πολύχρονων συζητήσεων επί το δύο αυτό φακέλου. Η επίδεξη συμφωνία θα δώσει όθηση στην εσωτερική αγορά μέσα από τον καθορισμό εναρμονισμένων κανόνων για την έγκριση τύπου και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και τη βελτιστοποίηση τη εποπτεία της αγοράς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Uh, so I'm going to, um, uh, invite members. Θα ήθελα τώρα οι βουλευτές να υποβάλουν ερωτήσεις επειδή έχετε έναν εκτενή κατάλογο αρμοδιοτήτων και θα συνεργαστούμε μαζί σας, έχουμε την κυρία Βερνιό και τον κύριο Κρέγ μαζί μας, τους δύο εισηγητές, σε σχέση με θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να λάβουν το λόγο οι δύο εισηγητές σε σχέση με τα πακέτα που έχουν αναλάβει και μετά τους εισηγητές, η κυρία Ρούλε θα λάβει το λόγο, ο κύριος Σβάμπ και άλλα μέλη που το επιθυμούν. Και η κυρία Πιέτη Κάινεν. Χαίρομαι που αναφερθήκατε και στη δική μου έκθεση για τα σκάφη αναψυχής. Η κυρία Βερνιό έχει το λόγο. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία για την παρουσία της και αρχίζοντας να κάνω ένα αστιάκι ίσως. Πολύ λίγοι συνάδελφοι είναι παρόντος. Και θα πω το εξή. Ίσως αυτή η συνάντηση, αν είχε γίνει στη Λευκοσία, θα είχε περισσότερους πιστούς, γιατί τουλάχιστον εσείς έχετε ήλιο. Τέλος πάντων, το λέω αυτά για να αισθανθούμε όλοι πιο άνετα. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Τώρα όσον αφορά τις δύο οδηγίες που μας απασχολούν στα πλαίσια της ενίας εσωτερικής αγοράς, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι αναφερθήκατε στις δημόσιες συμβάσεις, μιλήσατε στην αναλογία, στην ε, ποιότητα, αλλά άκουσα να λέτε επίσης ότι στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων θα ασχοληθείτε με το θέμα της μη τήρησης των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Και ιδιαίτερος είπατε ότι θα προσέξετε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ξέρουμε ότι είναι ο σκληρός πυρήνας της εσωτερικής αγοράς. Και συνεισφέρει όντως στην κοινωνική και στην εδαφική συνοχή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, που είναι ο δικό μου φάκελο, συμφωνούμε όλα τα θεσμικά όργανα στο ότι θα πρέπει όντω η κινητικότητα να βελτιωθεί, να δημιουργεί μεγαλύτερη ανάπτυξη, καλέ θέσει απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Είπετε όμως κάτι το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, δεδομένου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας και το δικό σας ως προεδρεύουσα χώρα και υπολογίζω στις προσπάθειές σας. Μιλήσατε για εμβάθυνση και βελτίωση εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη. Στην οδηγία αυτή είναι σημαντικό να παράσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες, να δείξουμε ότι η Ευρώπη έχει μια πραγματική προστιθέμενη αξία και να αφήσουμε στα κράτη περιθώριο δυνατοτήτων να ασκήσουν τις δικές τους αρμοδιότητες. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτή είναι η παρούσα δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε. Υπολογίζω λοιπόν σε εσά, διότι όπως είπατε ο πολίτης μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση από τα κράτη-μέλη. Στη χώρα μου δεν είναι εξαιρετικά τα πράγματα, ιδιαίτερα μάλιστα άσημα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προσφύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και την πράσιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών και θα κάνουμε πραγματικά, ε, θα δώσουμε τα σωστά μηνύματα για τη δημιουργία εμπιστοσύνης. Είσαστε μια μικρή χώρα μικρή προεδρία όπω λέμε, αλλά καμιά φορά οι μικρές προεδρίες κάνουν, αυτό πρέπει να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Γκρέσου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι από τη μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που βλέπω μια άλλη και νέα χώρα να προεδρεύει. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Εάν κρίνω την εμπειρία που δούμε μέχρι τώρα από την Κυπριακή Προεδρία, πρέπει να πω ότι όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μου φάκελο, επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό ιονός είναι αυτό για το μέλλον. Και αναφέρατε και κάτι άλλο. Είπατε ότι πιστεύετε στην ενιαία εσωτερική αγορά για τους πολίτες πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, θα ήθελα να μην υπάρχει πληθώρα προτεραιοτήτων στην ατζέντα σας και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι κάπως αρνητικό. Το πρόβλημά μου και ερώτησή μου είναι η εξής. Θέλουμε ε, να φτιάξουμε καλύτερη την εσωτερική αγορά. Δεν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάτε το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο πρέπει κάτι να κάνετε για να το πείσετε. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν ποια είναι η στρατηγική σας. Πώς θα προσπαθήσετε να ξεπεράσετε τα εμπόδια που υπάρχουν στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε πραγματικά να φτιάξουμε αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις πρώτα απ' όλα κύριε Υπουργέ. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ε κυρία Βερνάουτ. Να πω ότι ε, σε ό,τι αφορά ε, και για τα καλά της λόγια, να πω σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Εμείς ακριβώς θέλουμε να, να βλέπουμε όλες τις πτυχές του θέματος. Δηλαδή, πέραν από τη δυνατότητα πρόσβασης των μικρών μεσιών επιχειρήσεων, την όθηση στην ανάπτυξη, ε, θέλουμε να, ε, να δίνεται όθηση ε, στην αηφόρο ανάπτυξη, στην καινοτομία, αλλά και στην εφαρμογή σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές πτυχές που σχεδίζονται βεβαίως με το αντικείμενο της εκάστοτης σύμβασης και έχει μεγάλη σημασία να, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και βεβαίως η προστασία μέσα από αυτή την εφαρμογή και των ίδιων των εργαζομένων. Ε, σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τα επαγγελματικά ε, προσόντα, ε, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, ένα, ε, είναι ένας δύσκολος φάκελος. Ε, ε, όλοι πιστεύουμε στην ανάγκη να υπάρχει κινητικότητα στην Ευρώπη και πραγματικά υπάρχει μέσα από τις ε, ε, διμερείς μας επαφές ε, με τα άλλα κράτη θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και να εξεύρουμε λύσεις στην πολυπλοκότητα των θεμάτων. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει απέναντι στα επαγγελματικά προσόντα να υπάρχει εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Και οι πολίτες πρέπει πρώτα και κύρια ήδη να γνωρίζουν ε, τα δικαιώματά τους. Όμως είναι αλήθεια ότι οι διαφορές που έχουμε στην Ευρώπη σωστή ό,τι αφορά ε, και τα θέματα εκπαίδευσης και τα θέματα κατάρτισης δυσκολεύουν ε, το να προχωρήσουν αυτή η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, άρα θεωρώ ότι η σύγκληση πρέπει να είναι και σε πολλούς άλλους τομείς. Όμως είναι αναγκαία να, να βρούμε διέξοδο, γιατί έτσι θα ενισχύσουμε από τη μια και την κινητικότητα στην Ευρώπη, αλλά και από την άλλη ε, θα βοηθήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ε, των πολιτών ε, της κάτι χώρας όταν ξέρουμε ότι τα επαγγελματικά προσόντα είναι κατηχρωμένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ η αναφορά που έχετε κάνει, κυρία Βερνά, έχετε δίκιο ότι σαν μικρή Προεδρία θα προσπαθήσουμε ε, και να στείλουμε και τα σωστά μηνύματα αλλά και να λειτουργήσουμε ενός ένας ε, αξιόπιστος διαμεσολαβητής. Στα ε, θέματα που έθεσε ο κύριο Κρέσ, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Νομίζω ότι ο κύριο Κρέσ, προερχόμενο από μια μικρή χώρα, καταλαβαίνει πόσες δυσκολίες υπάρχουν στα μικρά κράτη όταν ασκούν την Προεδρία, ειδικότερα όταν είναι λίγο των προσωπικών. όμω, θεωρώ ότι Έχουμε αρκετά καλό προσωπικό και μπορούμε ακριβώ να δουλέψουμε μέσα σε ε, πνεύμα συνεργασία. Ε, για να ξεπεράσουμε αναφερθήκετε στα εμπόδια. Εμεί ε, ω μικρέ χώρε έχουμε περισσότερο την ανάγκη να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη. Και περισσότερη Ευρώπη σημαίνει ολοκλήρωση τη ενία αγορά. Καταλαβαίνουμε ότι ε, υπάρχουν δυσκολίε στου Η προσπάθεια μα ω Προεδρία είναι όσο το δυνατόν περισσότερου φακέλου από την ενιαία πράξη αγορά ε, για την ενιαία αγορά, την πράξη 1 και ταυτόχρονα, όπω είπα και στην αγωγή μου ομιλία, να σπρώξουμε και είμαστε ευτυχεί γιατί υπάρχει κινητικότητα μέσα από την ανακοίνωση τη ε, Επιτροπή να υιοθετήσουμε συμπεράσματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα του Δεκεμβρίου για την ενιαία πράξη αγορά 2 και παράλληλα να προχωρήσουν αυτοί οι φακέλοι. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε, ε, όμως ε, ε, θεωρούμε ότι η συνεργασία μας και με την Επιτροπή αλλά ιδιαίτερα με το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει να βρούμε πολλές φορές καλύτερες λύσεις και στο Συμβούλιο που συμφωνώ μαζί σας σε αυτά τα θέματα ίσως εκεί να παρουσιάζονται και οι περισσότερες δυσκολίες. Και βεβαίως υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να μορυγνήσουμε ώστε να, ε, να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση στην υλοποίηση των μέτρων για την νέα αγορά. Δεν φτάνει να εγκρίνουμε νομοθετήματα, πρέπει να παρακολουθούμε και στην πράξη το πώ υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, so the next two speakers... Ευχαριστούμε. Οι επόμενοι δύο ομιλητές είναι η κυρία Ρούλε και ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Καταρχήν για την παρουσία σας σήμερα εδώ, αλλά και για την παρουσίαση που μας κάνατε, για τα σημεία τα οποία υπογραμμίσατε και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Κυπριακή Προεδρία. Έχω δύο παρατηρήσεις και θα ήθελα ενδεχομένως να ακολουθήσει κάποια συζήτηση από αυτών των θεμάτων. Ανακοινώσατε στα σημεία τα οποία θέλετε να αποτελέσουν επίκεντρο της Προεδρίας σας, ε, σημεία τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι το Δεκέμβριο. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των δημόσιων συμβάσεων και Πιστεύω ότι ενδεχομένως θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά την πραγματική επίτευξη στόχων. Ίσως δηλαδή θα πρέπει για να φτάσουμε σε πραγματική απλοποίηση, σε νομική ασφάλεια, να πάμε λίγο πιο αργά έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πραγματικές, ε, πραγματική πρόοδο. Υπάρχουν ε, τομείς ε, οι οποίοι όπως ξέρετε δεν είναι εύκολο να περάσουν. Πληθώρα τροπολογιών έχουν υποβληθεί, συζήτηση σε αρκετά έντονο ε, τόνο έχει ήδη υπάρξει και βεβαίως το θέμα της συμφωνίας στην πρώτη ανάγνωση θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η Προεδρία σας για το θέμα αυτό. Η Δανέζικη Προεδρία, από ό,τι καταλάβαμε, δεν ε, είχε διαπιστώσει μεγάλη ομοφωνία για το θέμα αυτό. Εσείς τι έχετε να πείτε. Και δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ε, εκχώρησης ε, για θέματα υπηρεσιών. Είναι κάτι που σαφώς και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Προτιμούμε και σε αυτό το τομέα να υπάρξει συμφωνία να υπάρξει σωστή νομοθετική ρύθμιση και ενδεχομένω περισσότερο χρόνο αν αυτό είναι απαραίτητο. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το μεσημέρι συζητήσαμε για κάποια από αυτά τα θέματα και ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Άσχετο τώρα ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου το θέμα της ενιαίας αγοράς ε, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει είτε θέλουμε είτε όχι. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Επιτρόπου Μπαρνιά για τα θέματα εσωτερικής αγοράς. Ξέρουμε ότι θέλετε να κλείσετε, να ολοκληρώσετε κάποια συγκεκριμένα θέματα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Αναρωτιέμαι μήπως εδώ θα πρέπει για κάποια θέματα να κοιτάξουμε πολύ περισσότερο την ποιότητα και να μην βιαστούμε. Και βεβαίως ε, θα σας αναφέρω ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να δημιουργεί πολλές δυσκολίες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Εσείς λοιπόν εδώ εκπροσωπείτε μια προεδρία η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να την υποψιαστεί ότι βρίσκεται πίσω από κάποια συμφέροντα μεγάλων κρατών. Εσείς λοιπόν πραγματικά είστε υπέρ της ανάπτυξης και σίγουρα υπέρ περισσότερης διαφάνειας. Θα θέλαμε λοιπόν η συζήτηση για το πώς υλοποιούν παραδείγματος χάρη τα κράτη-μέλη την νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, για τις δημόσιες συμβάσεις, για το πώς υλοποιούν τα κράτη-μέλη την κοινοτική νομοθεσία γενικότερα. Εδώ θα θέλαμε μια μεγάλη συζήτηση και βεβαίως σε καμία περίπτωση αυτό το θέμα δεν πρόκειται να λυθεί έτσι εύκολα και να ξεπεραστεί έτσι εύκολα, αλλά υπάρχουν σήμερα προβλήματα υλοποίησης, υπάρχουν προβλήματα πνεύματος, αν θέλετε, των νομοθετικών κυμάτων και πολλές φορές βλέπουμε οδηγίες, οδηγίες κοινοτικές, οι οποίες δεν υλοποιούνται, ενώ το περιεχόμενό τους είναι πραγματικά αυτονόητο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στους δύο συναδέλφους. Ε, σε ό,τι αφορά το ε, ερώτημα της κυρίας Ρούτε, ε, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και γνωρίζω για την πληθώρα τροπολογιών που μπαίνουν στα θέματα δημοσίου συμβάσεων. Ε, και μιλούμε για πολλά ζητήματα, γι' αυτό στην απάντηση προηγούμενο μίλησα για πολλέ πτυχέ που αφορούν περιλαμβανοντικέ, κοινωνικέ πτυχέ. Όμω αυτό καμιά φορά ο ρυθμό ε, δεν καθορίζεται μόνο ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Εάν υπάρχουν συγκλήσει, εάν όλοι νιώθουμε την ανάγκη ότι αυτό ειδικότερα σε μια περίοδο που υπάρχει οικονομική κρίση στην Ευρώπη και χρειάζεται να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη χωρίς να παραβλέπονται βεβαίω ούτε όλες οι άλλε πτυχέ, είναι αυτό που πολλές φορές η ίδια ζωή που μας καθορίζει το ρυθμό ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα χωρίς να παραβλέπουμε βεβαίω ε, την ουσία του θέματος. Ε, και αυτό που μπορώ να διαβίωσω ω Κυπριακή Προεδρία ότι ε, στη βάση και αυτό που είπα στην προηγούμενη μου απάντηση θα προσπαθήσουμε να υπάρξει ουσιαστική ε, πρόοδος σε ό,τι αφορά ε, αυτούς τους ε, φαγγέλους. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα διαφορετικές και μεγάλες διαφορετικές απόψεις γύρω από τη συζήτηση του θέματος. Τώρα, στα θέματα της εκχώρησης των υπηρεσιών, να πω ότι είναι σημαντικό ε, να πούμε ότι οι υπηρεσίες είναι ένας σημαντικός τομέας ε, στην, ε, στην Ευρώπη και θα πρέπει ακριβώς μέσα από, τα, από αυτές αυτά τα νομοθετήματα να δώσουμε όθηση σε αυτόν τον σημαντικό τομέα που πιστεύω ότι σε πάρα πολλά ζητήματα είναι σημαντικός στην ίδια την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ίδια την οικονομία της. Στα θέματα που έθεσε ο, ο, Ανδρέας, ο, κύριος Ανδρέας Βάπη, να πω ότι ε, ε, και εδώ είναι παρόμοιο το, το ζήτημα γύρω από την ποιότητα και τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και η θέση του να μην βιαστούν Επειδή έκανε αναφορά στα, στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ε, ένα θέμα που συζήτησα εκτεταμένα ε, το πρωί στην ε, Επιτροπή Νομικών την Τζούρι. κοιτάξτε, εδώ δεν νομίζω ότι στα θέματα των δημιουργών της τεχνίας βιαστήκαμε. Νομίζω πήρε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ανεξάρτητο καμιά φορά ε, η, ταχύτητα που κινόμαστε από το εκεί που γίνεται ένας συμβιβασμός. Γιατί υπάρχουν τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ε, εκεί έγινε ένας συμβιβασμός που ε, δεν ικανοποιεί το Κοινοβούλιο, όμως ε, όπως είπα και το πρωί στη Τζούρι, ακόμα και στα θέματα που δεν είναι συνηθισμένα, να, που ακολουθείτε, μπορεί να ακολουθήσουμε μια συνήθιστη πρακτική παρέκκλησης από τη συνήθιη διαδικασία εάν πραγματικά υπάρχει η πολιτική βούληση και από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο να βρούμε λύσεις. Και είναι αυτό που τοποθετήθηκα και στο προεστικούριο ότι θεωρώ ότι ε, μπορούμε να βρούμε λύση. Ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα της, ε, που έθεσε για την υλοποίηση των νομοθεσιών, συμφωνώ. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Εγκρίνομαι και θέλουμε να εγκρίνουμε συνεχώς νέες οδηγίες, νέα νομοθετήματα που αφορούν την εσωτερική αγορά. Και ναι, υπάρχει ένα θέμα και συμφωνώ με τον κύριο Σβάπη πώς ε, παρακολουθούμε την υλοποίηση αυτών των νομοθετημάτων. Και όντως σε πάρα πολλά κρατημέλη υπάρχουν προβλήματα. Και είναι εδώ που πρέπει να, να συζητήσουμε ε, και να μπορέσουμε να είμαστε ε, να βρούμε μηχανισμούς όχι μόνο παρακολούθησης θα έλεγα καλύτερης επιβολής της, της εφαρμογής των νομοθετημάτων ε, στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Uh, um, ο κύριος Κοφεράτη για την επόμενη ερώτηση και ο κύριος Ζουβέ. Μιλούσαμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Ίσως θα μπορούσατε να μας ε, μιλήσετε για τη δική σας έκθεση ως προς τις εκχωρήσεις. Ο κύριος Κοφεράτη πρώτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των δημόσιων συμβάσεων. Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο Υπουργός, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες γιατί η κρίση, όπως γνωρίζετε, πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ουδής αποκλείεται. και δυστυχώς έχουμε ανησυχητικούς δείκτες ανεργίας και φτώχειας, κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και στη σχέση θεσμικών οργάνων και πολιτών. Νομίζω ότι υποτιμούμε τους κινδύνους που ενδεχομένως απορρέουν από αυτή τη ρήξη Εάν οι πολίτες θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, τότε θα μπορέσουν να αντιδράσουν διαφορετικά. Θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις δημοκρατικές αρχές και να απαρνηθούν αυτή τη σχέση με τα θεσμικά όργανα. Αυτό μπορεί να απορρέει είτε από τους φόβους είτε από τις ηλικέ δυσχέρειες. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Μιλάμε για ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά παράλληλα θα πρέπει να βρούμε εν χρόνο και λύσεις για τα προβλήματα φτώχειας και αποκλεισμού. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα και μας το υπενθυμίσατε και εσείς. Υπ' αυτή την έννοια, οι δημόσιες συμβάσεις είναι το, το σημαντικότερο όργανο που διαθέτουμε σύμφωνα με τον μηχανισμό του Keynes. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει, έχουν γίνει πολλές και ζωηρές συζητήσεις. Χρειάζονται, χρειάζεται μια στήριξη αυτού του σχήματος και θα πρέπει να υπάρχουν και συνοδευτικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει νομιμότητα και διαφάνεια. Δεν έχουμε ένα εναλλακτικό σχήμα από αυτή την κεινσιανική πολιτική για να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οργανωμένη εγκληματικότητα εκεί όπου διενεργούνται έρευνες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ σοβαρά πώς ε, προωθούνται αυτές οι συμβάσεις και πώς ε, ε, λειτουργεί το οικονομικό μας σύστημα μέσα στα πλαίσια του θεσμικού αυτού σχηματισμού. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Um, uh, uh, Πρόεδρος. είπα και ανέφερα ότι θα πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού. Πρόκειται για ένα νέο σχηματισμό του Συμβουλίου και μιλώντας με άλλους υπουργούς, πρώην υπουργούς, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει παρουσία όλων, διότι δεν υπάρχει υπουργό ανταγωνισμού σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση αυτά που είπε και ο κύριος Κοφεράτη και την ατζέντα ανάπτυξης, την αναπτυξιακή ατζέντα, ίσως θα πρέπει να μας μιλήσετε για μια συλλογική στρατηγική ανάπτυξης. Και πάντα υπάρχει η ευκαιρία για τους υπουργούς να συζητήσουν για μια πολιτική γενικότερα μέσα στα πλαίσια των επισήμων συμβουλίων. Όταν συνεργαζόμαστε με τις προεδρίες, μιλάμε για θέματα λεπτομερίας, αλλά όχι για θέματα προσανατολισμού των πολιτικών μας. Με βάση αυτά που είπε ο κύριος Κοφεράτη, μπορείτε να μας πείτε μερικά από τα μυστικά σας, δηλαδή τι έχει τεθεί επιτάπητο στο οποίο μπορεί να ενδιαφέρει και εμάς, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να ξεκινήσω από μια ε, διαπίστωση του κύριου Κοφεράτη και ευχαριστώ που το αναφέρει αυτό. Η κρίση αγγίζει όλες τις χώρες, όλα τα κράτη-μέλη. Ε, δεν πρέπει να δίνεται εντύπωση, ακόμα και στα κράτη-μέλη που σήμερα μπορεί να μην είναι εμφανές η κρίση, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε ε, προβλήματα στην κρίση. Ε, είναι δεδομένο, είμαστε δεμένοι σε μια ενιαία αγορά και γι' αυτό τα προβλήματα που αφορούν την ανεργία και τη φτώχεια ε, είναι φανή σήμερα ε, σε πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ότι το ανάφερα και σε άλλες περιπτώσεις ότι χαίρομαι γιατί η συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη επανέρχεται στην Ευρώπη. Το να περιοριστούμε μόνο σε πολιτικές ε, δημοσιονομικών κανόνων και περικοπών. Αυτό ε, πολλές φορές ε, και το είδαμε να εμφανίζεται σε μερικές χώρες, δημιουργά τα αντίθετα αποτελέσματα. Δημιουργά περισσότερη ύφεση, ενισχύει την αναργία και είναι γι' αυτό που είναι σημαντικό μέσα από τις οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο για ε, να τονώσουμε την αγορά, να δώσουμε ιδιαίτερα ε, δυνατότητες μέσα από την απλοποίηση και το διαδικασίο, ε, μέσα από τη διαφάνεια της παρέμβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι λέμε και είναι γεγονός αυτό το πράγμα γιατί είναι η πραγματικότητα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης. Ε, πρέπει να τους δώσουμε και είναι μέσα από την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη θα αντιμετωπίσουμε την ύφεση και μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούνται και περισσότερες θέσει εργασίας ε, για να αντιμετωπίσουμε την εργασία. Άρα ε, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο οι δημόσιες συμβάσεις για την ανάπτυξη αλλά και να δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα ε, να ε, υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, αλλά ειδικότερα να δραστηριοποιηθούν περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Στα θέματα που θέσε ο κ. Πρόεδρος, είναι αλήθεια ότι ε, ναι, ε, στο σχήμα, πρώτα πρώτα να πω ότι έχουμε στα υπόψη μα πω πρέπει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ε, και το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα, Ήδη με τη Γραμματεία του Συμβουλίου συζητούμε κάποια πράγματα που αφορούν τις διαδικασίες. Τώρα, βεβαίω, το πώ είναι ο υπουργό σε κάθε χώρα, αυτά τα αντιλαμβανόμαστε. Τώρα αναφέρεστε και σε ένα υπουργό, κύριε Πρόεδρε, που έχει πάρα πολλά κάτω από την αρμοδιότητα του. Όμω, ε, σε ό,τι αφορά την την ατζέντα, είναι θέματα βεβαίω που θα τα συζητήσω και με, ε, αύριο με την Επιτροπή Νίτρε. Ε, Πρώτα-πρώτα είμαστε στην Προεδρία μας, έχουμε θέσει ως προτεραιότητες την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας τη νεανική επιχειρηματικότητα, της επιχειρηματικότητα ε, ε, των γυναικών, τη δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς του επιχειρηματίε, τους έντιμου επιχειρηματίε που οδηγήθηκαν ε, σε πτώκευση. Να πω ότι αυτά θα είναι και αντικείμενο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας που θα, γίνει, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο στις 19 Ιουλίου ε, και η πρόθεση μας είναι να εκδώσουμε ε, συμπεράσματα στο τέλος του χρόνου. Άλλο ζήτημα που θέλουμε βεβαίω να προωθήσουμε είναι τα θέματα βιομηχανικής πολιτικής και εδώ αναμένουμε από την Επιτροπή την έκδοση ανακοίνωση για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε και εδώ στην έκδοση συμπερασμάτων. Είναι πολιτικές που θα μας στρέψουν και στην πραγματική οικονομία που το έχει αρκετή ανάγκη σήμερα η Ευρώπη, δηλαδή τη στροφή στην πραγματική οικονομία για να οθεί ε, όθηση ε, στην ανάπτυξη αλλά και στον ανταγωνισμό της ίδιας ε, την ίδιων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και τέλος βεβαίως είναι και το πρόγραμμα COSME το οποίο θα συζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση του πριν από τέλος του 2012. Ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, ήθελα να αναφέρω ζητήματα ακριβώς που ε, ε, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα μας βοηθήσουν πραγματικά να επαναφέρουμε την ευρωπαϊκή οικονομία στο δρόμο της ανάπτυξης. Well, thank you very Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας ε, ενδιέφερε ιδιαίτερα το άτυπο αυτό συμβούλιο το οποίο μας είπατε ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα γίνουν πολλά σχόλια μέσα στα πλαίσια των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει να κρατήσετε και εσείς στεναρή στάση εναντί των ΜΜΕ. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση το τι ακριβώς κάνατε σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, σε σχέση με την ηλεκτρονική πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Ο κύριος Ζουβέν ίσως έχει να μας πει μερικά πράγματα για το θέμα των εκχωρήσεων που μας απασχολεί ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των δημόσιων συμβάσεων τον έπεισα να μας πει μερικά πράγματα. Έχουν γίνει πολλές έρευνες και αναζητήσεις και εάν άλλοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις προς τον Υπουργό, είναι και η τελευταία σας ευκαιρία. Καταρχήν είναι το λόγο στον κύριο Ζουβέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ διότι μας αφιερώνετε τον πολύτιμο χρόνο σας και μας πρέπει να πω ότι χαιρετίζω την γνώση των διαφόρων φακέλων. Φαίνεται από τις απαντήσεις που λέτε. Τώρα, όσον αφορά τις διάφορες συμβάσεις παραχώρησης. Θελήσει η Επιτροπή να υπάρχει η κατάλληλη νομοθετική πράξη ώστε να μπορεί κανείς ε, να νομοθετεί για θέματα συμβάσεων παραχωρήσεων για έργα και υπηρεσίες. Μέχρι τώρα είχαμε για τις εργασίες οδηγία και δεύτερον για τις υπηρεσίες λέγαμε ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του δικαίου και τελικά πρέπει να πω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ενεργός νομοθεσία επί τα τελευταία, νομολογία με συγχωρεί τα τελευταία δέκα χρόνια, άρα είναι σωστό αυτό που θα γίνει. Αναφέρατε τις δημόσιες αγορές πρώτα απ' όλα και δεύτερον τις παραχωρήσεις. Και τις παραχωρήσεις, τις συμβάσεις παραχωρήσεων, θέθηκαν κάποια ερωτηματικά και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο γενικότερα, διότι σχεδόν ομόφωνα, και εγώ ως εισηγητής το γνωρίζω πολύ καλά, θεωρούμε ότι στο κείμενο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότητες των παραχωρήσεων κάνει λοιπόν μια δημόσια αγορά κατά κάποιο τρόπο την ε, παραχώρηση. Το λέω συνοπτικά. Μας φάνηκε ότι το κείμενο είναι πολύπλοκο, δίσκαμπτο στις διαδικασίες που προβλέπει και εγώ το κείμενο το οποίο είχα την τιμή να υποβάλω στο Κοινοβούλιο πριν από κάποιες μέρες και το οποίο είναι στη θέσή σας, προσπαθεί να τονίσει τις ιδιαιτερότητες των συμβάσεων παραχωρήσεων που είναι κάποιες ατελείς συμβάσεις, όπως λέγουν οι νομικοί, δηλαδή συμβάσεις οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν στον χρόνο. Στην ε, μελέτη που έγινε και στη Γαλλία και στη Νότια Αμερική, απεδείχθη ότι δύο χρόνια μετά την υπογραφή τους αυτές οι συμβάσεις αναθεωρούνται. Στις ε, δημόσιες συμβάσεις έχουμε μία δισκαμψία, ενώ στις συμβάσεις παραχωρήσεων Πρέπει να έχουμε μία ευληξία, ευληξία μία καμψία. Το κείμενό μου, λοιπόν, προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα κριτήρια ευελιξίας. Επιμένω λοιπόν, δεδομένου ότι εσείς τώρα θα ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, ότι θα πρέπει αυτό το νομοθετικό ε, μέσον που θεωρείται ως ε, προσέγγιση light να μπορέσει στις δημόσιες αρχές να δώσει κάποια εξουσία την οποία θα διατηρήσουν κατά τη διάρκεια όλων των διαπραγματεύσεων για να γίνει ευέλικτο αυτό το μέσο. Πρέπει να πω ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε πριν από δύο χρόνια και θα κάνουμε σφάλμα εάν θα πρέπει αυτές τις συμβάσεις παραχωρήσεων να τις ε, συμπεριλάβουμε γενικότερα σε αυτά τα οποία θα πούμε για τις ε, δημόσιες αγορές. Διότι νομίζω ότι θα αφαιρέσουμε αυτό το στοιχείο. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας και εμείς θα να το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Πολύ χρήσιμα ήταν αυτά τα σχόλια. Θα ζητήσω από τον Υπουργό να σχολιάσει. Αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ε, ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ, κύριε Ζωβίν. Να πω ότι ε, έχετε δίκιο, θα πρέπει να τις δούμε διαφορετικά ε, τις συμβάσεις παραχώρησης από τις, ε, συμβάσεις, ε, τις δημόσιες συμβάσεις της αγοράς. Εμείς θα πω μια γενικότερη θέση ως Προεδρία. Θεωρούμε ότι είναι σωστό ότι ε, μια απλοποιημένη μορφή οδηγία ε, με περιορισμένους κανόνες ε, που θα διασφαλίζουν όμως τις αρχές της ε, διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης θα συμβάλλει στην ειδοποίηση και ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων και αυτό έχει να κάνει με την ανάκαψη και την μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή. Πρέπει να μεριμνήσουμε ακριβώς στην ορθή διαχείριση αυτών των δημοσίων συμβάσεων. Είναι μια προσπάθεια που ε, χρειάζεται να υπάρξει βεβαίω μια ισορροπία γιατί από τη μια θέλουμε να δώσουμε ενώθηση ε, στον ανταγωνισμό αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε από την άλλη ότι χρειάζεται διαφάνεια και ορθή ε, διαχείριση σε ό,τι αφορά τι ε, συμβάσει ε, παραχώρηση. Και είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτή την κατεύθυνση, ε, μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει που θα κινηθούμε ως ε, Προεδρία. Well, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε, που μας αφιερώσετε τόσο χρόνο σήμερα το απόγευμα και με τους ε, συντονιστές και το Προεδρείο γευματίσαμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Μας εντυπωσίασε όταν ήρθαμε να σας δούμε το ότι έχετε μια πολύ ισχυρή ομάδα που χειρίζεται πολύ καλά όλους τους φακέλους, φαίνεται ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και πραγματικά βλέπουμε ότι έχετε αναλάβει δεσμεύσεις σοβαρές με αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν την πράξη για την ενιαία αγορά και την ενιαία αγορά ε, γενικότερα. Η πράξη αυτή πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο Θέλουμε επίσης να υλοποιηθεί. Υπενθυμίζω την έκθεση του κυρίου Γκρέχ του 2010, την νέα αγορά για τους πολίτες και τους καταναλωτές. Χαιρόμαστε λοιπόν που εσείς συνεχίζετε προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει και το ψήφισμα το οποίο τον Ιούνιο υιοθετήσαμε στο Στρασβούργο και στο οποίο ε, εκθέτουμε τις ιδέες μας για το νέο, ε, για το σύνολο μέτρων όταν θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα στον επόμενο γύρο. Έχετε λοιπόν την πλήρη υποστήριξή μας για να υλοποιήσετε αυτή την πάρα πολύ φιλόδοξη ατζέντα που έχετε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει, είναι θέμα Υψηλή προτεραιότητας, φαίνεται από όλε τις συζητήσει. Πιστεύω επίσης ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την επίσκεψή μα στην Κύπρο είδαμε ότι εμείς συνειδητοποιείται πλήρως τη σημασία των ΜΜΕ για την εικόνα. Νομίζω ότι μπορείτε με την εμπειρία που έχετε να διαδραματίσετε ηγετικό ρόλο και στα θέματα των δημοσίων συμβάσεων δείχνετε τι μπορεί να γίνει, διότι εδώ ε, παρέχουν υπηρεσίες και στον τομέα αυτό πάρα πολλές μιμιές στην οικονομία σας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό για όλη την Ευρώπη, για όλες τις οικονομίες. Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά. Χαίρομαι που είναι εδώ πολλά μέλη της ομάδας σας που σας υποστηρίζουν. Τα γνωρίζουμε σιγά σιγά όλα τα άτομα που σας ε, συνοδεύουν. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ελπίζουμε ότι κατά τη προεδρία θα μπορέσουμε να σας ξαναεπισκεφθούμε στην Κύπρο και ξέρω ότι με έχετε συμπεριλάβει στην διάσκεψη που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου για με την ολοκλήρωση της ε, εβδομάδας της ε, τουρκικής αγοράς και ίσως και κάποια άλλα δύο-τρία μέλη θα θελήσουν να έρθουν κάποια στιγμή να δούνε και εκπροσώπους των ΜΜΕ της χώρας σας. Υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσει, Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να τι αντιμετωπίσουμε το επόμενο εξάμεινο. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία και ελπίζουμε ότι και στο μεταξύ διάστημα θα μπορέσουμε να σας ξανασυντήσουμε. Ελπίζουμε ότι θα ξαναεπισκεφτείτε και πάλι την Επιτροπή μας στο τέλος της Προεδρίας σας για να μας μιλήσετε για τις επιτεύξεις σας. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την επισκεψή σας σήμερα το απόγευμα. το гориστό

Uh, so, colleagues, um, uh, Αποχαιρέτησα τον Υπουργό και σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στη συζήτηση. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Κυπριακή Προεδρία. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ντένις Ντεγιόγκ, που είναι ο εισηγητής για θέματα προϋπολογισμού και θα μας μιλήσει για το σχέδιο γνωμοδότησης. Στη συνέχεια έχουμε και μερικούς σκιώδεις. Ο κύριος Σβάμπ, είσαστε σκιώδη στη θέση του κυρίου Βαντεκάμπ. Α, όχι, ο κύριος Βαντεκάμπ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μπουσόη, η κυρία Ρούλε είναι εδώ. Άλλοι είναι παρόντες, άλλοι απόντες. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Jong να μας παρουσιάσει τη νομοδότηση. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας. Ο κύριος Jong έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Μάλκομ. Πραγματικά υπάρχουν ε, κάποιες τροπολογίες τις οποίες βεβαίως θα σας παρουσιάσω και θα ενημερώσω και τα μέλη της Επιτροπής. Η γνωμοδότηση η οποία παρουσιάζει την περίοδο λιτότητας που έχει επιπτώσεις για όλους μας δεν μπορεί να αγνοηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν εδώ μία κριτική προσέγγιση. Είχαμε αρκετές συζητήσεις με τους υπαλλήλους της Επιτροπής καθότι θα πρέπει να γίνει διαφορά, διαφοροποίηση μεταξύ των κεντρικών hardcore δραστηριοτήτων, αυτών δηλαδή που θεωρούμε εμείς σημαντικές και αυτές που θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο πιο δευτερεύουσες παραδείγματο χάρη σεμινάρια κατάρτισης ή διάφορα άλλα γεγονότα τα οποία οργανώνονται και όταν συζητήσαμε με υψηλά ιστάμενους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώσαμε ότι και οι ίδιοι δεν ξέρουν ακριβώς ποιο θα είναι το περιεχόμενο όλων αυτών των διοργανώσεων αλλά ε, τις έχουν παρόλα αυτά προβλέψει μπας και χρειαστεί όπως μας είπαν. Θα θέλαμε λοιπόν πραγματικά να να προβλεφθεί το ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για όλες τις δραστηριότητες τυποποίησης. Η τυποποίηση είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε. Η δημόσιες αρχές θα πρέπει παραδείγματος χάρη να βοηθήσουν να στηρίξουν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ε, την διαδικασία τυποποίησης έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν και αναρωτιέμαι εδώ αν θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε την νομοθεσία από την τυποποίηση. Η τυποποίηση είναι κάτι πραγματικά που αφορά τον ιδιωτικό τομέα και υπάρχει και μία χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, η οποία είναι κάτι το τελείως διαφορετικό σε σχέση με την νομοθεσία. Άρα εδώ μπορεί σαφώς και να υπάρξει και μία εξοικονόμηση πόρων. Δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο, το Solvit. Όπως ξέρετε, συμπεριλαμβάνεται το Solvit σαν ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτοντάς τον με τα αρχικά προς υπόμνηση. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το Solvit. Υπάρχει το Solvit, υπάρχει το Europe Advice και άλλες οδηγίες πλαίσιο, οι οποίες πρώτον είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, και εάν προβλεφθεί ένας προϋπολογισμός για τις τρεις-τέσσερις αυτές οδηγίες, καταλαβαίνετε ότι η Επιτροπή αποκτά τη δυνατότητα να δείξει ότι διαχειρίζεται με πολύ καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, τα θέματα αυτά. Πρόκειται λοιπόν για ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι λιτός και εμείς σαν Επιτροπή έχουμε τις δικές μας ε, προτεραιότητες. Για τα πιλωτικά προγράμματα, όπως παραδείγματος το χάρη το Φόρουμ για την ενιαία αγορά. Πρόκειται για μία εκδήλωση που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και μόλις ακούσαμε τον ε, Υπουργό όσον αφορά την ε, μείωση της συχνότητας αυτής της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Okay. Thank very much. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ρεαλιστική αυτή η αξιολόγηση. Θα δούμε. Ο κύριος Φαμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί να είναι παρόν ο σκιώδης εισηγητής, αλλά σίγουρα θα είχε ακούσει με το ίδιο ενδιαφέρον ε, την παρουσίαση του ε, εισηγητή μας, με το ίδιο ενδιαφέρον ε, που την άκουσα και εγώ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι για τα σημεία από το 1 έως το 7 καταρχήν συμφωνούμε και εκεί που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την άποψή μου όσον αφορά τις προτεραιότητες βεβαίως αυτών των σημείων αν και βεβαίως εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για τα μέσα που θα διατεθούν για αυτές εδώ τις δαπάνες. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για θέματα Ευρωπαίων πολιτών εσωτερικής αγοράς και εκεί πραγματικά ε, πρέπει να θέσουμε όλο το βάρος της προσοχής μας. Το σημείο 2, εκεί που αναφέρεται το εξωτερικό προσωπικό, ε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις προτάσεις. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε τις προτάσεις στους, ε, στους υπόλοιπους ε, τομείς. Όσον αφορά την αποθήκευση, εδώ πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Κατά τα άλλα, σύμφωνο με αυτά που μας είπε ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τις εκτιμήσεις που έγιναν και τις παρατηρήσεις για την έκθεση De Jong. Κάποιες συστάσεις λοιπόν έκανε με λογική και με σωστά επιχειρήματα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε όπως λέτε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο λιτότητας και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να την μετατρέψουμε σε περίοδο ανάπτυξης. Η ΙΜΚΟ νομίζω ότι έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, διότι πρέπει να βελτιώσει την ενιαία εσωτερική αγορά και να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για να λειτουργήσει σωστά ε, και κάθε παραγωγικό τομέα και να βελτιωθεί η κατάσταση των καταναλωτών. Οτιδήποτε κάνουμε λοιπόν θα είναι πάρα πολύ θετικό για να περάσουμε από την λιτότητα στην ανάπτυξη. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω την δυνατότητα να κάνουμε και κάποιες υποδείξεις σε σχέση με το κείμενο που μας παρουσιάστηκε για να δούμε με ποιο τρόπο ο προϋπολογισμός του 2013 μπορεί να ενισχύσει από την οπτική γωνία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς δράσεις αποτελεσματικές κατά της ανεργίας των νέων, φερρυπίν, υπέρ της δημιουργίας κινήτρων για την απασχόληση και την ανάπτυξη, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες, το κράτος δηλαδή, τις διάφορες χώρες μέλη να βελτιωθούν και η ανταγωνιστικότητα επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και τελικά θα ήθελα να προσθέσω ότι οι διάφορες υποδείξεις που θα κάνουμε θα πρέπει να στοχεύουν στο ότι η υποδημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς δεν θα ξεχάσει ποτέ και το κοινωνικό σκέλος. Διότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μία εύρωστη ενιαία εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουζόη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, δουλειά που επιτέλεσε, για αυτή την πολύ σημαντική ομοδότηση. Υπάρχουν πολλές ιδέες με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα, υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες τις οποίες θα πρέπει κάπως να συζητήσουμε και να έχουμε και κάποιες διευκρινήσεις. Όπως ήδη είπαν και οι προλαλήσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα και κυρίως τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε το εξή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περικοπές αυτομάτως και στον κοινοτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο κοινοτικό προπολογισμό υποστηρίζει την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη σε περιοχέ όπου τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δαπανίσουν περισσότερα χρήματα και κυρίω σε περιοχέ στι οποίε από κοινού μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στο σημείο 3 λέει ο ότι στην γραμμή 02, 03, 01 θα πρέπει να θέσουμε τις κατάλληλες προτεραιότητες. Σωστά το λέει, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες. Διότι συμφωνώ απολύτως ότι θα ήταν καλύτερα να κάνουμε καλύτερα κάποια πράγματα με λιγότερα κονδύλια, αλλά θα πρέπει να δούμε και στην πράξη μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Πρέπει να πω ότι ως πρώην εισηγητής ε, εγώ απογοητεύομαι, διότι η Επιτροπή για το Solvit φέτο και για την ενιαία ιστορική αγορά δεν προβλέπει ε, δεσμεύσεις κονδυλίων για να βοηθηθεί η αγορά. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ θα καταθέσω τροπολογία για αυτό το θέμα καθώς και για τον προπολογισμό. Και τελειώνοντας θα πω ότι υπάρχει πρόταση από, τον, ε, από την συνάδελφη Ρόζα Τούν για την εσωτερική αγορά να αναλάβουμε μία προπαρασκευαστική δράση για το φόρουμ και θυμάστε το πρώτο φόρουμ το οποίο έγινε στην Κρακοβία στην οποία συμμετείχαμε κάποιοι και ήταν επιτυχία ελπίζουμε να οργανωθεί περαιτέρω ένα φόρουμ που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο την νησθενία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ η κυρία Ρούλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι συμμερίζουμε απόλυτα παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν. Θα πρέπει όντω αυτά το χρόνο τη οικονομική δυσκολία να προσέξουμε πάρα πολύ πώ να πανούμε τα κονδύλια που διαθέτουμε. Και θα πρέπει τα ποσά τα οποία δίδονται για, από τον κοινοτικό προορισμό για κάποια project να είναι χρήσιμα. Θα ήθελα να πω το εξή τον κύριο Ντογιόγκ. Δεν είναι πάντα πάρα πολύ ακριβή όσον αφορά τι δαπάνε τη Οικομισιόν, όσον αφορά του διαφόρου φακέλου. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ακούσουμε και την ίδια την Επιτροπή με μεγαλύτερη ακρίβεια για να μα πει τι πρεσβεύει στα διάφορα σημεία. Όταν αφορά το Solvit, είναι πολύ πιο παλιό θέμα. Πάντα το χειριζόμαστε κάπως βιαστικά. Θα πρέπει να επανέλθουμε. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος De Jong, θα πρέπει για κάποια θέματα να μας δώσει πιο πολλές εξηγήσεις η Επιτροπή. Θέλουμε η Επιτροπή να ενθαρρύνει την συμμετοχή των ΜΜΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων που εκπροσωπούν την κοινωνία, αλλά θα θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μας πει με ακρίβεια περί τίνος πρόκειται. Όσον αφορά την πράξη για την ενιαία αγορά, συμφωνώ με τη Ρόζα Τούν, όπως και ο κύριος Μπουζόη, πιστεύω ότι όντως ήταν μια πραγματική επιτυχία και θα πρέπει μια τέτοια δράση να τη συνεχίσουμε. Για τους Ευρωπαίους πολίτες η εσωτερική αγορά δεν είναι ακόμη η πραγματικότητα και μεταξύ των πολιτών υπάρχει ένας κάποιος σκεπτικισμός όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ποιες είναι οι επικρίσεις που γίνονται και οι φόβοι που εκφράζονται. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω. Συμφωνώ με τη γενική υποστήριξη του θέματος. Γιατί νομίζω ότι είναι ρεαλιστική και λογική πρόταση. Χρειάζεται βεβαίως να δούμε τους δελφικούς χρησμούς αυτής της πρότασης. Δηλαδή υπάρχουν ε, πολλά, πολλές αμφιγνωμίες και πολλές αμφισημίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ποιες ε, είναι επακριβώς οι προτεραιότητες που ορίζουμε. Ο Ντένις λέει στο άρθρο 7 ότι η πολιτική υπέρ των καταναλωτών είναι απόλυτη η προτεραιότητα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές την πολιτική των καταναλωτών κατά όλων των άλλων. Φυσικά θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους καταναλωτές, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό μας ε, μέλημα θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ενώσεις καταναλωτών στα νέα κράτη-μέλη, εκεί που υπάρχουν πιο αδύναμοι οργανισμοί και φορείς. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης, εκφράσατε το σκεπτικισμό σας σε σχέση με τις γραμμές του προϋπολογισμού για προγράμματα κατάρτισης. Αυτό θα πρέπει ίσως να το πούμε πιο, ίσως θα πρέπει να φέρουμε πιο καθαρά. Ως προς το θέμα της τυποποίησης, καθίσταται σαφές ότι έχουμε ορίσει προτεραιότητες για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ. Είναι θέματα τα οποία θα τα εντάξουμε ευρύτερα στις επενδύσεις για την τυποποίηση και νομίζω ότι ως προς το θέμα των ε, συμβουλευτικών οργανώσεων μας ενδιαφέρει να ε, λάβουμε υπόψη ιστοσελίδες που σχετίζονται και με τις επιχειρήσεις αλλά και με τους καταναλωτές. Εκεί όπου υπάρχουν σημεία διεπαφής και να προωθήσουμε μία ενιαία πύλη έτσι ώστε να εξορθολογήσουμε και να προβούμε σε οικονομίες. Εδώ θα πρέπει κάπως να συμπιέσουμε τον προϋπολογισμό για να προωθηθεί αυτός ο εξορθολογισμός κατά καλύτερο τρόπο και να συμβαδίζει με αυτά που προαναφέραμε. Ως προς τον προϋπολογισμό για τα τελωνία, κυρία Λεγκρίπ θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις και γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη, δεν ανταποκρίθηκαν στις ε, δεσμεύσεις τους έτσι ώστε να εξευρεθούν πόροι για να προωθηθούν τα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα των ε, τελωνίων και του εξορθολογισμού της λειτουργίας τους, ιδιαίτερα ως προς τις μεγάλες δαπάνες. Αυτό θα είναι ένα σημείο εκκίνησης σε σχέση με διοργάνωση σεμιναρίων, σεμιναρίων, αν μιλάμε για την εφαρμογή των νέων συστημάτων, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να περικόψουμε σε αυτούς τους τομείς, γιατί αν δεν υπάρχει κατάρτιση, τότε δεν βελτιστοποιείται η επένδυση που γίνεται στο νέο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να επιτελεστεί αρκετή εργασία, αλλά θίξατε πολλά ουσιώδη ζητήματα. Υπάρχουν άλλα μέλη που θα ήθελα να λάβουν το λόγο πριν ε, λάβει το λόγο ο Ντένις. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει εκπρόσωπος από την Κομισιόν, από τις υπηρεσίες της Κομισιόν που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Όλοι είσαστε με κατεβασμένο το κεφάλι. Δεν θέλετε να υπερασπιστείτε στον προπολογισμό σας. Θα δούμε τι θα κάνουμε με το επόμενο στάδιο εργασιών. Ντένις, έχεις το λόγο. Έχεις ένα χρονοδιάγραμμα. Θέλεις να συνοψίσεις και να μας ε, μιλήσεις και για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχω και εγώ μπροστά μου. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σαφής για τις προθέσεις μας ως προς τις τροπολογίες αυτές, γιατί θέλω να δώσουμε μεγαλύτερο περιεχόμενο στη γνωμοδότηση. Το θέμα αυτό το είχαμε συζητήσει με την Κομισιόν και μαζί με τη Γραμματεία και τώρα που ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γνωρίζουμε πού μπορούμε να κάνουμε περικοπές και που όχι. Αναφέρομαι στην παράγραφο 3 και θα επανέλθω σε αυτή. Σε σχέση με την τυποποίηση, Εάν το συζητήσετε με την Κομισιόν, βλέπετε ότι πολλά από τα χρήματα ε, τοποθετούνται εκεί που θέλει η ΙΜΚΟ, δηλαδή τη συμμετοχή των ε, ΜΜΕ και των καταναλωτών στη διαδικασία τυποποίησης. Υπ' αυτή την έννοια Νομίζω ότι έχει, έχουν γίνει πολλές περικοπές στον τομέα της τυποποίησης της τάξης των 5 εκατομμυρίων. Η Γενική Διεύθυνση της Αγοράς τόνισε ότι δεν μπόρεσε να καταδείξει πού υπάρχει προστιθέμενη αξία, εάν υπάρχει. Και Ίσως θα γινόταν μείωση κατά 1,5 εκατομμύριο χωρίς να υπάρχει, αρνητική, να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στην αγορά. Ως προς τα τελωνία, το Συμβούλιο θέλει να μειώσει κατά 5-6 εκατομμύρια. Δραστικές μειώσεις λοιπόν προβάλλει, οι συζητήσεις συνεχίζονται και θα επανέλθουμε στο ζήτημα. Ως προς την παράγραφο 3, για τις δαπάνες βλέπουμε ότι είναι υψηλότερες από την ε, περσινή χρονιά. Έγιναν αρκετές συζητήσεις με την σχετική γενική διεύθυνση και βλέπουμε πώς μπορούν να γίνουν ε, περικοπές. Δηλαδή, εκεί όπου πραγματικά δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία θα πρέπει να μειώνονται οι δαπάνες. Σε σχέση με το Solvit θα γίνει μια μείωση της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Χρειάζεται εξορθολογισμός και θα πρέπει να περιορίσουμε τις κεφαλίδες του προϋπολογισμού ως προς τα επιμέρους ε, ζητήματα, αλλά το Solvit στοιχίζει χρήματα και γι' αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το κεφάλαιο. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο επί του παρόντος και θα, θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Ως προς τα γενικότερα σχόλια, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προβούμε σε επιμέρους διευθετήσεις και νομίζω ότι η ενιαία αγορά έχει μεγάλη σημασία για τις απασχολήσεις και την ανάπτυξη. Αυτό θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε στη γνωμοδότηση. Φυσικά χρειάζονται περικοπές, αλλά η ενιαία αγορά θα πρέπει να προωθηθεί μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών μας ρυθμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρονοδιάγραμμα. Βλέπω μπροστά μου ότι θα πρέπει να ορίσουμε την υποβολή τροπολογιών στις 27 Ιουλίου για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην Επιτροπή Υπολογισμών που θα ε, ψηφίσει στις 3-4 Οκτωβρίου. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 6 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή και θα ψηφίσουμε επίσης στις 6. Είναι η πρώτη εβδομάδα που θα συνεδριάσουμε μετά την πράσινη εβδομάδα. Και στις 6 του μηνός θα ε, συνεδριάσουμε. Στις 21 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το κοινό κείμενο με τους προϋπολογισμούς. Βεβαίως ε, συνεργαστήκατε με τη Γραμματεία και θα πρέπει να υποβάλλετε τις τροπολογίες γιατί πολλοί θα λείπουμε στη Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα Γι' αυτό θα σας διαβιβάσουμε τις σκέψεις μας από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Λοιπόν, από τις 3 μέχρι 6.30 στις 3 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες σας. Στις 6, με συγχωρείτε. Τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες της έκθεσης Ρόιτοβα ε, είμαστε δύο λεπτά πριν θα πρότεινα να αρχίσουμε ακριβώς στις 5 παρατέταρτο γιατί πολλοί δεν έχουν έρθει και θα ήθελα η κυρία Ρόιτοβα να μας εξηγήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας. Και αυτό θα είναι και το τελευταίο θέμα μας, οι ψηφοφορίες. Και μετά θα προχωρήσουμε στους συντονιστές.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

Uh, Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχουν έλθει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Καλό θα ήταν να είσαστε και λίγο περισσότεροι προηγουμένω. Ήταν ο Υπουργό ε, στις 3 η ώρα, ο Προεδρεύων. Η κυρία Ρούλα ήταν μόνο εδώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέχουμε ώστε όταν έρχεται κάποιος υπουργό να είμαστε λίγο περισσότερο στην άθεση. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά καλύτερα θέλω να είστε κάπως περισσότεροι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ψηφοφορίες για τις εκθέσεις της κυρίας Ρόιτοβα. Πρόκειται για ασυνήθη ψηφοφορία, διότι έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν οριζοντίως όλες τις οδηγίες. Θα ήθελα να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις, αν θέλει, για τον τρόπο τον οποίο θα ψηφίσουν και τα κάποια στιγμή που υπάρχουν. Η κυρία Ρότα, να αρχίσουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι μαζί με τη γραμματεία προετοιμάσαμε με τέτοιο τρόπο τους καταλόγους ψηφοφορίας, ώστε όλες οι αλλαγές οριζόντιας μορφής που αφορούν όλες τις οδηγίες να ψηφιστούν στην πρώτη οδηγία που αφορά την πρώτη έκθεση Επαναλαμβάνω λοιπόν όλες τις οριζόντιες θα τις ψηφίσουμε στην πρώτη έκθεση και μετά θα ψηφίσουμε όλες τις άλλες. Επίσης πρέπει να πω ότι έχετε τον τελικό κατάλογο ψηφοφοριών. Και για τους επισκέπτες, στο βάθος της αίθουσας έχουμε μία άλλη εκδοχή. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Όποιος λοιπόν πάρει το κείμενο από το βάθος της αίθουσα, υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει, κατα... δεν, υπάρχει... δεν είναι παρεμφερής ο κατάλογος των ψηφοφοριών. Αλλά των συναδέλφων οι φάκελοι δεν έχουν λάθη. Έχετε το λόγο και πάλι, Πρόεδρε. Υπάρχει κάποια σύγχυση. Έχουν του κόκκινους φακέλους οι συνάδελφοι του ΕΛΚ. Οι σοσιαλιστές τους έχουν. Τέλος πάντων. Να διευκρινίσουμε δύο πράγματα πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα, ξέρω ότι κάνατε στα τεχνικά θέματα πάρα πολλή δουλειά. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο τομείς μπορούμε να ψηφίσουμε on block διότι υπάρχουν θέματα που μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. Μπορείτε λοιπόν να μου πείτε πού μπορούμε να ψηφίσουμε, σε ποια κομμάτια on block. Δεύτερον, ξέρω ότι η κυρία Βανβεοντιού ήθελε να παρουσιάσει κάποια νέα στοιχεία, αλλά από όσο καταλαβαίνω, μετά από τη σημερινή συζήτηση, την πρωινή συζήτηση, είπαμε ότι κάποιες τροπολογίες θα αποσυρθούν από εδώ, και αργότερα θα επανέλθουν όταν θα γίνει πλήρης αναθεώρηση όλων των οδηγιών. Ας μου κάνει ε, σήμα λοιπόν η κυρία Βερδιού κάθε φορά που υπάρχει κάποια τέτοια μικρό αλλαγή. Λοιπόν, για να αρχίσουμε. Ε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλά προβλήματα ψηφοφορία, αλλά κρατήστε και τις κάρτες σας. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα. Εναρμόνιση των επιθεσιών σχετικά με τη διάθεση των αγορά πλών δοχείων πίεση. Τροπολογία 3 τη εισηγητρία. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 5. 6 και 7 μπορούμε να τι ψηφίσουμε μπλοκ. Ναι. 5, 6 και 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 και 9 μπορούμε να τι ναι. ψηφίσουμε μαζί. Πολύ καλά, υπέρ, κατά, δεν θα αναφέρω τις αποχές, αν κάποιος θέλει να απόσχει να μου το πει. Λοιπόν, συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, συμβιβαστική 2, εγκρίνεται και πάλι. 14 και 15 μαζί, όχι 16 λέει η κυρία Λοιπόν, 14 και 15, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Ίσως πρώτα απ' όλα Ελέγξτε αν λειτουργούν οι κάρτες σας. Την 16 ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 20. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Εδώ οι 42, 43, 44, 45, 46, 47 και 48 αφορούν έτοιμα πιστοποίησης από ανεξάρτητους οργανισμούς. Η Κομισιό είναι παρούσα μήπως. Εάν κατάλαβα καλά, η Κομισιόν προσωπικά στην συνάντηση αυτή πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση να κάνει μελέτη επιπτώσεων. Περί αυτού δεν πρόκειται Κριστέλ. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα προβλήματα αυτά πιστοποίησης. Δεν ξέρω αν θέλει να λάβει το λόγο. Διαφορετικά θα αποσύρω όλες αυτές τις τροπολογίες που μου φαίνεται παρόλα αυτά ότι για την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια ότι είναι σημαντικές. Αλλά αν υπάρξει δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής, την εμπιστεύομαι. Κομισιόν είναι παρούσα, μήπως. Παρακαλώ. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό, αλλά ίσως θα ήταν χρήσιμο. Ναι, Σήμερα το πρωί η κυρία Μπρίγκμαν είπε ότι το 2013 θα γίνει μια ευρεία κλίμακος διαβούλευση για όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο που φορά τα βιομηχανικά προϊόντα και θα εξετάσουμε τα προβλήματα και τα θέματα τα οποία στα πλαίσια αυτής της άσκησης που το κάνουμε θα πρέπει να επιλύσουμε. Σήμερα το πρωί ανέφερε κάποια εισαγωγές που αφορούν προσωπικής χρήση προϊόντα από τρίτες χώρες και γι' αυτό αν τα πλαίσια αυτή τη διαβούλευση αυτά τα θέματα μπορούμε να τα καλύψουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ο σωστό τρόπο να το χειριστούμε είναι αυτός βεβαίω. Λοιπόν, οι επόμενε τροπολογίε. 21, 22, 23, 24 μπορούν να ψηφιστούν μαζί. 21, 22, 23, 49, 25, 26, όχι την 24, όλες αυτές τις 6 on block. Υπέρ κατά εγκρίνονται. Στην επόμενη σελίδα έχουμε την... Ε, όχι, στο κάτω μέρος σελίδας. 27, 28, υπέρ κατά εγκρίνεται. 50, υπέρ κατά Απορρίπτεται. 29, 30 μαζί. Μπορώ. Όχι. Μόνο την 29. 29. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30. Ποιος είναι υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 17 προς 12. 33, 31, 33. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία, εγκρίνεται. 31, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά εγκρίνεται 34 υπέρ κατά εγκρίνεται τώρα φτάνουμε στην στις ε, αιτιολογική ε, σκέψη το 4 συμβιβαστική 6 συμβιβαστική εγκρίνεται ε, τροπολογία 2 της κυρίας Ρόιτοβα εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με Ομοφωνία 21 μελών. Συγχαρητήρια κυρία Ρόιτοβα. Στο τέλος. Στο τέλος, για να μην χάνουμε χρόνο, θα σας συγχαρούμε για όλες τι εκθέσεις. Επόμενη έκθεση. Όργανα ζήγησης μη αυτόματης λειτουργίας. Έχετε το ίδια σελίδα με μένα, 31-32. Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 33 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 35 της κυρίας Βερνιό. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. απορρίπτεται. Ω προσθήκη 34 τη κυρία Ρότοβα, υπέρ κατά εγκρίνεται. On block τώρα. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Αποσύρεται η 5. Ψηφίζουμε την 43. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 44 αρχίζει η ψηφοφορία όλοι είστε κατά εντάξει απορρίπτεται λοιπόν 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53 και 54. On block. Υπέρ. Κατά εγκρίνονται. 49. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 7. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αποσύρεται η 9, 55, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 20. Μία απορρίπτεται 28 εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά εγκρίνεται, 67, 68, 70, 72, on block, υπέρ, ε, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, απορρίπτονται και 29, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για την αναδιατύπωση, ε, σχετικά με τα όργανα ζήγησης μη αυτόματης λειτουργίας. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. 28 υπερψήφισαν. Περνούμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Αναδιατύπωση για την διαθεσιμότητα στην αγορά και τον των ενεργητικών ειρών εμπορικής χρήσης. Αρχίζουμε με την 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται χωριστή ψηφοφορία στην 33 της κυρίας Βερνιό μπορείτε να δείτε που χωρίζονται την ψηφίζουμε λοιπόν χωριστά δεν θα τη διαβάσω τώρα το πρώτο μέρος ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 6. Ρόιτοβα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, 10. Εγκρίνεται επίσης. Μπορούμε να ψηφίσουμε την 34, ε, 35 και 36 μαζί. Όχι την 36. 34 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία, απορρίπτεται. 35 υπέρ. υπέρ κατά απορρίπτεται 36 απορρίπτεται επίσης 14 εγκρίνεται 39 εγκρίνεται 46 εγκρίνεται 29 και 30 μαζί. Και 48. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση του συνόλου του ψηφίσματος. Αρχίζει η ψηφοφορία για τις εκρηκτικές ύλες. Λίγη ψηφοφορία και εγκρίνεται η έκθεση αυτή με 27 ψήφους υπέρ και καμία κατά. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. 4. Πρόκειται για τα συστήματα προστασίας για ιδιαίτερα εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Αυτό δεν ισχύει εδώ στην Επιτροπή μας βέβαια. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε όλα on block. Νομίζω ότι υπάρχει μια πρόταση να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Δεν υπάρχει κανείς που είναι κατά. Ωραία. 29, 30, 14, 15, 36, 26. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται όλες οι τροπολογίες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για ιδιαίτερα εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 28 υπέρ και κανείς κατά. Και τώρα θα μιλήσουμε για το επόμενο θέμα της ημερησίας. Είμαστε στο 28. Να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 29 και 40. Κατά. Εγκρίνονται. Και τώρα... Α, νομίζω ότι κάποιοι ήταν κατά. 41 υπέρ, κατά. 41, ξαναψηφίζουμε, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 43, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται 44, υπέρ. 6, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 45 καταπίπτει, 46 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 47 υπέρ, ε, κατά, εγκρίνεται, 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα να τα ψηφίσουμε unblock, όχι το 48. 48. 48 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Για ποια άλλη τροπολογία θέλετε ξεχωριστή. 24. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν 11, 12,

όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται όλες. Επόμενη σελίδα όλες τις υπόλοιπες μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί 32, 33, 70, 71, 72 υπέρ κατά εγκρίνονται όλες και τώρα είμαστε σε αιτιολογικές σκέψεις. Ένα. Τροπολογία ένα. Υπέρ. Κατά. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35 καταπίπτει. 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το όλο κείμενο. Ψηφίζουμε. 27 υπέρ, μία αποχή, κανείς κατά. Ωραία. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο θέμα, ηλεκτρολογικός υλικός που προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης και εδώ πρόκειται για διατύπωση. 10, 12, 14 μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Και τώρα έχουμε 17, 18, 29, 31, 32 και το σημείο 28 υπέρ κατά. Εγκρίνονται όλες μαζί. Οι επόμενες μπορούν να ψηφιστούν μαζί. 16, 18, 23, 47, 48, 49. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Συμβαστικές 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Η 1, η 5 και η 40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 26 υπέρ, κανείς κατά. Το επόμενο σημείο, έχουμε άλλα δύο, ε. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα είναι το επόμενο θέμα. Να ψηφίσουμε on block, όλα μαζί. Ωραία. Και προφορικές και όλα. Α, ε, έχετε ήδη πάει διακοπές εσείς. Πολύ ευχαριστώ να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες on block. Ναι. Υπέρ λοιπόν. Όλες οι τροπολογίες ψηφίζουμε. Κατά. Ωραία. Όλες εγκρίνονται. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου. Υπέρ. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Τέλος της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, κανείς κατά. Κυρία Ρόιτοβα, αξίζετε συγχαρητηρίων. Uh, uh, Πραγματικά ήταν δύσκολο το έργο σας, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Ρόιτοβα, πριν διακόψουμε. Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι τα χειροκροτήματα που άκουσα πρέπει να πάνε πραγματικά στον βοηθό μου. Uh, comment? Η Επιτροπή θέλει να πει κάτι όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα. Okay. Ωραία. Είναι και το τελευταίο θέμα για σήμερα. <coughs> Κυρίες και κύριοι, τελειώνει με το θέμα αυτό η ημερήσια διάταξη. Θα ακολουθήσει η συνάντηση των ε, συντονιστών, η οποία μπορεί να αρχίσει αμέσως. Σας ε, υπενθυμίζω ότι θα συνεδριάσουμε <coughs> στις 6 Σεπτεμβρίου, 5η, στις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και σας εύχομαι καλές διακοπές. Ξέρω ότι δεν θα πάτε βέβαια διακοπές, θα εργάζεστε όλο τον Αύγουστο και ελπίζω να σας δω ξεκούραστος το Σεπτέμβριο. Τέλος της συνεδρίασης και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Olympics reception. Mrs. McClarkin is inviting you to the Olympic Games reception at 6 o'clock. Is it 6 o'clock, Emma? Phil.